Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, uh, σας παρακαλώ πολύ, όποιος δεν θέλει να μείνει για τις επεξηγήσεις ψήφων, να αποχωρήσει από το ημικύκλιο, ώστε να μπορέσουν όσοι ενδιαφέρονται για τις επεξηγήσεις ψήφου να τις παρουσιάσουν χωρίς καθυστέρηση. Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος δεν θέλει να μείνει για τις επεξηγήσεις να εγκαταλείψει την αίθουσα της Ολομέλειας σε ένδειξη συμβασμού προς τους συναδέλφους που πάλι θέλουν να κάνουν επεξηγήσεις ψήφου αλλά και να προλάβουν το αεροπλάνο τους. Thank Σας ευχαριστώ. Επεξηγήσεις λοιπόν. εγγύηση